κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίσω την έναρξη των εργασιών μας. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής για την